Αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί μας προσκεκλημένοι, παρακαλώ καθίστε. Αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στο δεύτερο τμήμα της σημερινής ημέρας για τα online μαθήματα, την ανώτερη εκπαίδευση και την ηλεκτρονική μάθηση. Θα ακούσουμε πρώτα την κυρία Γκρέιν Κόνολ από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ στο Ηνωμένο Βασίλειο και αμέσως μετά θα έχουμε μία συζήτηση στο πάνελ. Οι ερωτήσεις θα ακολουθήσουν τη συζήτηση του πάνελ. Δεν θα γίνουν αμέσως μετά την παρουσίαση της ε, κυρίας Κόνολ. Και μία ανακοίνωση για τους διερμηνείς. Στη διάρκεια της παρουσίας της κυρίας Κόνολ θα παρακολουθήσουμε ένα σύντομο βίντεο, μια σύντομη βιντεοτενία που φυσικά δεν χρειάζεται να την ε, μεταφράσατε. Αυτά, ευχαριστώ και ο λόγος στην κυρία Κόνολ. Good morning. It's a pleasure. Καλημέρα σα, Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Είναι μάλιστα ηλιόλουστη η μέρα σήμερα στι Βρυξέλλε. Εγώ θα σα δώσω μια εικόνα στα επόμενα 30 λεπτά περίπου για την ε, ηλεκτρονική μάθηση ω τομέα και ως τι, αυτό, τι συνέπειση έχει αυτό για την ανώτατη εκπαίδευση. Θα ξεκινήσω δίνοντα σα ε, μια χρονική γραμμή των βασικών οροσίμων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 20-30 ετών και έπειτα θα δούμε κάποιες τεχνολογικές τάσεις για το μέλλον. Εγώ θα σας αναφέρω κάποιες, υπάρχουν πολλές που μπορώ να σας αναφέρω, κάποιες βασικές τάσεις. Και στη συνέχεια θα δούμε ένα από τα συστήματα κλειδιά που έχουμε ως θεσμοί για να στηρίξουμε τους μαθητευόμενους, στα συστήματα διαχείρισης μάθησης δηλαδή. Και έπειτα θα σας μιλήσω για ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα παράδοξο σχήμα ότι παρά την πληθώρα τεχνολογικών ε, μέσων που υπάρχουν δεν χρησιμοποιούνται εκτεταμένα γιατί οι δάσκαλοι δεν έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες. Και θα σας περιγράψω τη δουλειά που κάνουμε τα τελευταία 10 χρόνια περίπου για να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε νέες προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό της εκμάθησης. Θα σας δείξω κάποια εργαλεία που έχουμε αναπτύξει και κάποια παραδείγματα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τεχνολογίες ώστε να προωθήσουν διάφορες προσεγγίσεις μάθησης και τέλος ε, θα σας δώσω κάποιες σκέψεις που μπορούν να προκαλέσουν ε, τη συζήτηση στο πάνελ. Στο 2007 μια ομάδα εξημών στον τομέα περίπου 30 ημών προσπαθήσαμε να ορίσουμε τι σημαίνει e-learning, ηλεκτρονική μάθηση και βασικά καταλήξαμε στον εξή ορισμό, ότι πρόκειται για την ανάπτυξη και την έρευνα τη εφαρμογή τεχνολογιών στην εκπαίδευση πολλές διαφορετικές λέξεις έχουν χρησιμοποιηθεί, δηλαδή τεχνόλογοι στην ε, παιδεία, δίκτυο, βελτίωση των ε, τεχνικών, Τη εκπαίδευση μέσω τεχνολογιών. Εγώ θα μείνω στο e-learning, στην ηλεκτρονική μάθηση, γιατί στην ουσία ε, περιέχει όλα αυτά. Την δεκαετία του 80 άρχισα, εγώ να ασχολούμαι με αυτό τον ε, τομέα και ε, τότε αναδύθηκαν τα πρώτα μέσα για ε, εργαλεία όπως το Toolbook ή Authorware που μπορούσε κανείς να αγοράσει δηλαδή κάποιες ε, κασέτες εκμάθησης και μετά ε, εμφανίστηκε το ίντερνετ, το διαδίκτυο και είδαμε διάφορα συστήματα διαχείρισης ε, όπως το Rule, ε, Blackboard και τα λοιπά. Μετά είχαμε τις κινητές συσκευές, είχα ένα φίλο που έκανε δακτορικό στις κινητές συσκευές πριν ε, να ξαπλωθούν τόσο πολύ. Θυμάστε κάποια πρώτα κινητά τηλέφωνα που ήταν τεράστια και ξαφνικά ολόκληρο το δακτορικό του ήταν για τα σκουπίδια λόγω της δημιουργίας αυτών των νέων εργαλειών. Μετά είχαμε τη δημιουργία των ε, παιχνιδιών και ε, των ανοιχτών ε, εκπαιδευτικών πόρων όπου το ανοιχτό πανεπιστήμιο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το MIT, άρχισαν τα, συστήματα, τα ανοιχτά συστήματα εκμάθησης. Μετά είδαμε τα κοινωνικά μέσα, ο Τίμο Ράιλι, ε, φίβρε την ε, λέξη web tool το 2003-2004 και στη συνέχεια είδαμε τα ηλεκτρονικά βιβλία και τις συσκευές αυτές όπως το iPad όπου μεταμορφών μεταμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο διαβάζω, χαζεύω στο ίντερνετ και τέλος είδαμε την μαζική ανάδεση ανοιχτών μαθημάτων online όπου συχνά συμμετέχουν χιλιάδες χιλιάδων ε, άνθρωποι. Κάποιες λοιπόν από αυτές τις τεχνολογικές τάσεις και εδώ μιλώ για, τον, για την έκθεση την ετήσια σε σχέση με τις τεχνολογίες, όπου βλέπουμε ποιες θα είναι αντίκτυπος τεχνολογίας σε δύο-τρία χρόνια. Κάποιες από τις τάσεις που τονίζονται λοιπόν είναι τα κινητά και τα ηλεκτρονικά βιβλία, προσωπική εκμάθηση, έτσι από ενδιαφέρον. Πόσοι από εσάς έχετε iPad ή ταμπλέτα, εν πάση περιπτώσει, κάποιου είδους. Είναι εντυπωσιακό πόσος κόσμος ε, τα έχει, αυτά, τα έχει αυτές τις συσκευέ. προσωποποιημένη ε, μάθηση, ατομική μάθηση, ώστε ο καθένας από εμά να μπορεί να διαλέξει ένα συγκεκριμένο είδο εργαλείων και προτιμήσεις για να μάθει πόσοι αγαπούν το Facebook, πόσοι μισούν το Facebook θα έπαιρνε ώρα να το συζητήσουμε. Έχω δύο παιδιά, το μεγαλύτερό μου μισή. Μισή το Facebook. Θεωρεί ότι είναι διαβολικό εργαλείο, ότι εγώ είμαι μανιακή. Έχουμε λοιπόν πολύ διαφορετικές ε, απόψεις. Τώρα, ε, το, οι υπολογιστές και το σύννεφο, τι μπορεί να υπάρχει στο σύννεφο ορισμένοι ας πούμε στέλνουν το email τους στο σύννεφο Τώρα, πανταχού παρούσα μάθηση. Αναμένουμε να είμαστε online παντού και πάντα. Και στην ουσία νομίζουμε ότι θα μείνουμε άπρακτοι αν δεν έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ. Μετά έχουμε την ιδέα του φέρε τη δική σου συσκευή. Αυτό το λαμβάνουμε υπόψη στις δομές μας για τους φοιτητές μας. Δηλαδή τα περιβάλλοντα είναι τεχνολογικά διευκολυμένα. Έχουμε αρκετές μπρίζε Το Wi-Fi μας είναι αρκετά καλό για να μπορεί να στηρίξει 200 φοιτητές που ταυτόχρονα θέλουν πρόσβαση στο ίντερνετ. Και έπειτα ε, ένα πολύ νέο καυτό θέμα είναι οι αναλύσεις της μάθησης. Αυτό σημαίνει ότι πέρα από τα συστήματα διαχείρισης της μάθησης υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν καλύτερα για το πώς διαδρούν οι φοιτητές μας online, να δούμε πού εντοπίζουν τα προβλήματά τους και να τους βοηθήσουμε. Πού και πού επίσης ε, συναντώ κάτι που δείχνει εδώ ε, κάτι το τελείωσε τρελό που θα αλλάξει τελείως. Σας δείχνω μια στιγμή αυτό το βίντεο της Google. Yeah. Um, meet me in front of Strand Books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 agree. That's pretty Ελπίζω ότι συμφωνείτε πως είναι πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά. Εγώ βέβαια δεν θα ήθελα να φοράω τέτοιου είδους γυαλιά όταν οδηγώ, αλλά σίγουρα τέτοιου είδους ε, πράγματα έχουν τεράστιο δυναμικό για την εκπαίδευση και πρωτότυπα αυτών των συσκευών υπάρχουν πλέον. Για να επανέλθουμε τώρα στην ουσία των, της τεχνολογίας, για να δούμε πώς μπορούν να στηρίξουν τους ε, μαθητές μας. Ε, έχουμε λοιπόν κάποια συστήματα διαχείρισης ε, της μάθησης και μόλις τελειώνω ένα ενημερωτικό έγγραφο της UNESCO που θα είναι διαθέσιμο στο site της UNESCO τους επόμενους μήνες, όπου εγώ... Αναφέρω τα διάφορα συστήματα τεχνολογικά που είναι διαθέσιμα στα διάφορα ε, ε, ιδρύματα και τι, από τι ακριβώς αποτελούνται. Πέρα από το Blackboard, Sakai και το Null υπάρχουν διάφορα συστήματα διαχείρισης, αλλά βασικά μπορούμε να τα μοιράσουμε σε έξι είδη. Πρώτον, δημιουργία περιεχομένου. Για παράδειγμα, στο Blackboard μπορεί κανείς να φορτώσει κείμενα πολύ μέσα κτλ. Μπορεί να το ομοδοποιήσει σε φακέλους ή να τα έχει σε ένα πρότυπο διαρθρωμένο. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία επικοινωνίας όπως τα φόρουμ συζήτησης μέχρι ε, εργαλεία για παρουσίαση, blogs, εργαλεία συνεργασίας όπως το Wikis, κάποια συστήματα μάθησης έχουν και ε, συνδέσεις για οπτικοακουστικές ε, διασκέψεις, ε, μετά έχουμε μέσα αξιολόγησης, ε, δηλαδή χαρτοφυλάκια και ηλεκτρονικά, διευκολύνσεις φόρτωσης για τους φοιτητές, εργαλεία φόρτωσης και έπειτα εργαλεία ανείχνευσης. Ε, αυτό το κεντρικό σύστημα λοιπόν διαχείρισης της μάθησης οδηγεί στα σε άλλες λειτουργίες του Ιδρύματος, δηλαδή που κάνει τις αιτήσει του, που είναι τα μητρώα, τα αρχεία, οι πόροι για την, την, την ε, βιβλιοθήκη ή τα μητρώα τους, μέχρι δηλαδή την αποφύτισή τους. Βασικά αυτές είναι, αυτά είναι τα βήματα και τα εργαλεία. Θα ήθελα να κοιτάξουμε τα βασικά, δύο από τα βασικά εργαλεία μέσα στο σύστημα διαχείρισης της ε, μάθησης. Καταρχήν έχουμε τα διάφορα φόρουμ, τα διάφορα βήματα που δίνουν ένα δομημένο χώρο για μη συγχρονισμένη συζήτηση. Επειδή υπάρχει αυτή η χρονική υστέρηση, μπορεί να είναι πολύ καλά για να ενθαρρυνθεί ο προβληματισμό, η περισυλλογή, να χρησιμοποιηθούν για απαντήσει, αλλά και ω ένα άτυπο, ε, ένας άτυπος κοινωνικός χώρος. Εγώ έκανα δύο μαθήματα στο ανοιχτό πανεπιστήμιο online, μαθαίνοντα ισπανικά θα πρέπει να πω ότι όλα τα χρόνια που είμαι ερευνήτρια σε αυτόν τον τομέα, το να είμαι online φοιτήτρια ήταν πιο πολύτιμο από οποιαδήποτε έρευνα έχω κάνει, γιατί έτσι κατάλαβα πραγματικά ποια είναι τα ζητήματα του να είναι κανείς ε, μαθητής online. Και έχουμε ένα φόρουμ που χρησιμοποιούμε, δεν το συντόνιζε ο διδάσκαλο, ήταν πολύτιμο όμω το φόρουμ, μοιραστήκαμε πόρου. υπήρχε ένα φοιτητή τον οποίο όλοι μισούσαμε, Εμεί ήμασταν στη βδομάδα 4, εκείνο ήταν στη βδομάδα 12 και μα έδινε κάτι χάρτε του μυαλού που μα κάνουν όλου να ε, τσαντιζόμαστε φρικτά. Ε, Υπάρχουν blog που εξηγούν πώς ε, χρησιμοποιείται το κάθε φόρουμ. Ξέρω ότι δεν μπορείτε να διαβάσετε το διάγραμμα, αλλά υπάρχει ένα σύνδεσμος κάτω-κάτω. Υπάρχει επίσης ένα σύνδεσμος για το EduCause που περιγράφει τι είναι τα blogs και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Εκεί υπάρχει μια ολόκληρη σειρά τέτοιων ενημερωτικών σημειωμάτων για τις διάφορες τεχνολογίες. Είναι τα 7 πράγματα που πρέπει κανείς να ξέρει για τα blog, για τα wikis, για το πορτοφόλιο. Σας τα συστήνω. Βασικά το διάγραμμα αυτό είναι η χρήση των φοιτητών ή των, των διδασκάλων των blog, όταν συγγρα... συντάσσουν ή όταν διαβάζουν και σχολιάζουν κάτι. Έχουμε δηλαδή στην ουσία μια συλλογή προσωπικών συνδέσμων και σχολείων. Μπορεί κανείς να προσθέσει σχόλια και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ώστε να προωθήσει τον προβληματισμό κατά τη διάρκεια των ε, μαθημάτων. Όταν, για παράδειγμα, θέλει οι φοιτητέ να σκεφτούν τη θεωρία τους, ε, όταν, ας πούμε, σπουδάζουν για να γίνουν καθηγητές, δάσκαλοι, και μετά να δεις πώς θα το εφαρμόσω στην πράξη. Wikis, άλλη μια σύνδεση σε αυτό το διάγραμμα κάτω-κάτω, ένα σύνδεσμος που σας δείχνει πώς οι φοιτητέ και οι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Wikis. Είναι ένας χώρος για ομάδες και προωθεί την μη συγχρονισμένη συνεργασία αν κρατάς μητρό το τι έχει κάνει ο καθένας είναι ένας καλός χώρος για ομαδικές δραστηριότητες. Για να συγκρίνουμε τα τρία λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι τα φόρουμ συζήτηση είναι καλά για συντονισμένες συζητήσεις, επίλυση προβλημάτων, ερωταπαντήσεις, τα blogs είναι πολύ καλά για το προσωπικό προβληματισμό, ατομικό προβληματισμό και τα wikis είναι συνεργασία και ομαδική δουλειά. Αυτά είναι βασικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούνται στα συστήματα διαχείρισης της εκμάθησης. Θα μπορούσαμε να περάσουμε ένα πολύ χρόνο μιλώντας για όλες αυτές τις καταπληκτικές τεχνολογίες και το πώς ε, προωθούν διάφορα είδη μάθησης και θα επανέλθω αργότερα για να σας δώσω παραδείγματα συμπεριλαμβανομένων παραδειγμάτων για την εκμάθηση γλωσσών αλλά παρά το γεγονός ότι έχουμε αυτά τα εκπληκτικά εργαλεία για να προσφέρουμε στους μαθητές και στους δασκάλους σπουδαίους τρόπους για να επικοινωνούν και να συνεργάζονται και παρά το γεγονός ότι έχουμε ε, πολλούς, δωρεάν τέτοιους πόρους, ε, οτιδήποτε θέλουμε να γνωρίζουμε υπάρχει στο ίντερνετ. Οπότε τίθεται το ερώτημα, τι είναι, ποιος είναι ο ρόλος ενός επίσημου ιδρύματος όταν τα πάντα είναι δωρεάν και θα επανέλθω σε αυτό αργότερα παρά όλα αυτά δεν τα εκμεταλλευόμαστε πλήρως. Αντιθέτως, απλώς λίγο στην επιφάνεια έχουμε αγγίξει αυτόν, το, το δυναμικό αυτών των τεχνολογιών και μάλιστα πολύ συχνά επαναλαμβάνουμε κακή παιδαγωγική, κακές παιδαγωγικές μεθόδους, δηλαδή ξεφυλίζουμε βιαστικά το ίντερνετ. Οι δάσκαλοι συνήθως λένε ότι δεν έχουν χρόνο, αλλά ούτε και δεξιότητες για να τα εκμεταλλευτούν αυτά. Μήπως μιλάω πολύ γρήγορα, ρωτάει η ομιλήτρια. Ναι, εντάξει. Λίγο γρήγορα. Λίγο γρήγορα. Όχι, όχι. Αν αρχίσω να μιλάω πολύ γρήγορα, κάντε μου νόημα. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα, το κενό ανάμεσα στις δυνατότητες και στην πραγματικότητα της τεχνολογίας είναι αυτό που με απασχολεί στην έρευνά μου και έχουμε αναπτύξει μια νέα προσέγγιση για να σχεδιάσουμε εργαλεία για την εκμάθηση. Βοηθά αυτό τους δασκάλους να σκεφτούν από την εσωτερική πίστη που έχουν στην διδασκαλία με βάση την εμπειρία τους για διαλέξεις ή ε, εργαστηριακές ε, ε, δοκιμές σε πρακτική εφαρμογή και έτσι τη βάση την σχεδιάζουμε πιο ορτά και άρα πιο κατανοητά για τους υπόλοιπους. Ως δάσκαλοι ε, εστιαζόμαστε στην, στο περιεχόμενο ενώ αυτή η προσέγγιση θέλει να δώσει στο δάσκαλο να καταλάβει και να μοιραστεί τις δραστηριότητες που μπορεί να μοιραστεί μαζί του. Ε, μόλις υπέβαλα μια πρόταση για να δημιουργηθεί ένα βιβλίο, ένα, μια ανθολογία σχεδιασμού μάθησης, δηλαδή περιπτώσεις, περίπου 100 περιπτώσεις, 100 διαφορετικοί τρόποι να σκεφτεί κανείς το σχεδιασμό <coughs> της μάθησης. Και θα σας δείξω κάποιους από αυτούς. Καταρχήν, Έχουμε τρεις πτυχές ε, όσον αφορά την, το σχεδιασμό της μάθησης. Η καθοδήγηση, η οπτική του παρουσίαση και όχι το κείμενο μόνο και έπειτα η πρόθεση τρόπων για να μπορέσεις να, την, να μοιραστείς αυτή τη γνώση. Για να σχεδιάσεις το, την μάθηση μιας δραστηριότητας, καταρχήν πρέπει να έχουμε την πρακτική, τη διδακτική πρακτική, ε, το πώς πιστεύει ότι μεταδίδει τη γνώση του, έπειτα τα χαρακτηριστικά του μαθητή, ε, τα πολιτιστικά ζητήματα, τον τρόπο με τον οποίο θα διδάξει ας πούμε, Άγγλους ε, μαθητές που θα είναι διαφορετικός από ότι να διδάξεις φοιτητές στη Σιγκαπούρη και έπειτα διάφορες παιδαγωγικές προσεγγίσεις καθώς και τις τεχνολογίες και ποια χαρακτηριστικά προσφέρουν αυτές οι τεχνολογίες. Είναι επίσης σημαντικό να λάβει κανείς υπόψη και το θεσμικό πλαίσιο καθώς και τους εξωτερικούς παράγοντες. Πολλά θέματα λοιπόν καθορίζονται από τις επαγγελματικές προδιαγραφές. Ας πούμε, οι μηχανικοί πρέπει να ακολουθούν τα στάνταρ του σώματός της. Οι χημικοί ε, στη, στο Ηνωμένο Βασίλειο, α πούμε, πρέπει να επακούν την ε, Βασιλική Ακαδημία Χημικών, για παράδειγμα. Ένα θέμα είναι λοιπόν να δούμε τα χαρακτηριστικά του μαθήματος. Τι θέλουμε να περιλαμβάνει. Ε, μπορεί να ε, πρόκειται για κάποια μαθήματα συνεργασίας, να υπάρχουν παραδείγματα, αξιολογήσεις, εξετάσεις, ε, διαγωνίσματα. Πρέπει κανείς να καταγράψει τα στοιχεία που θα είναι μέσα στο μάθημα, μέσα στο υλικό και τα στοιχεία που δεν θα περιλαμβάνονται εκεί. Το έχουμε κάνει αυτό εκατοντάδε φορέ και είναι πολύ καλό να ξέρει ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι σχεδιασμού. Μετά, έχουμε ένα, επίσης ένα χάρτη του, να δείξουμε τι είδου στήριξη υπάρχει. Μπορεί να υπάρχουν στάνταρ σύνδεσμοι, μπορεί να υπάρχουν σύνδεσμοι που βοηθούν και στηρίζουν ενημέρωση για την ε, βιβλιοθήκη ή για δεξιότητες μελέτης, ε, τι είδους περιεχόμενο και εμπειρία αναμένουμε, τι είδους ε, προβληματισμό και επίδειξη. Για παράδειγμα, για τους μαθητές γλωσσών, στην αρχή μπορεί να κάνουμε ένα διαγνωστικό διαγώνισμα για να αξιολογήσουμε το επίπεδο γνώσεών τους και ούτω καθεξής. Να δούμε δηλαδή το, να καταγράψουμε το είδος του προβληματισμού και της επιδεξικέπητα, το, τη φύση της επικοινωνίας και της συνεργασίας στη διάρκεια του μαθήματος. Εδώ έχουμε αυτό που ονομάζεται προφίλ δραστηριότητας, όπου κανείς ε, καταγράφει ε, ρητά τι κάνουν οι μαθητές και πόσο χρόνο δαπανούν εδώ. Δηλαδή, να διαβάσουν κάποιο κείμενο, να δουν ένα βίντεο, να ακούσουν κάποιο podcast, να ε, χειριστούν πληροφορίες, επικοινωνικές δραστηριότητες, ας πούμε να συμμετέχουν σε ένα φόρουμ, παραγωγικές δραστηριότητες, να φτιάξουν ένα αρχιτεκτονικό μοντέλο, να φτιάξουν ένα δοκίμιο. Ε, πειραματικά θέματα, προσαρμοστικά, πολύ πιο ειδικευμένα. Πρόκειται για μόντελινγκ ή προσωμιώσεις. Μπορεί να έχει δηλαδή κανείς ένα εκρεμές και μπορεί ο φοιτητής να πρέπει να αλλάξει το, τη συχνότητα των ταλαντώσεων. <coughs> Επίσης, ε, αξιολόγηση. Θα πρέπει να δώσουν πόσο χρόνο ε, χρησιμοποιούν για να ανταποκριθούν σε αυτές τις δραστηριότητες. Ας πούμε, ε, το υλικό για την Ισπανία, για τα ισπανικά μάλλον ήταν πάρα πολύ, αλλά το δικό μου μικρότερο, ας πούμε, μικρότερη μου λίστα ήταν η λίστα της επικοινωνίας, επειδή ακόμα δεν είχα τις γνώσεις. Εδώ Έχουμε αξιολόγηση όλων αυτών, δεν πρόκειται να σας τα πω όλα αυτά με λεπτομέρειες. Όλες αυτές οι διαφάνειες υπάρχουν στην έντυπα που σας έχω δώσει. Αλλά βασικά ήταν πιο ελεύθερη, πιο δημιουργική, πιο διαφορετικός ο τρόπος. Ε, ε, ε, ο κόσμος δηλαδή έρχεται να σκέφτεται διαφορετικά τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζει την ε, μάθηση. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα από το Open University, το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Έχουμε ένα σύστημα πολλαπλών ερωτήσεων. Οι φοιτητές μπορούν να συνδεθούν και να πάρουν έτσι αρκετά λεπτομερείς αξιολογήσεις. Εδώ έχουμε επαναλήψεις ε, και πρακτική για τα ισπανικά, για παράδειγμα. Ε, μπορεί να κάνεις διάφορες ασκήσεις, να συνδεθείς με άλλους εγώ, ας πούμε, συνδέθηκα με μια Σκοτσέζα που επίσης μάθανε Ισπανικά. Κινητή μάθηση, οι κινητές συσκευέ έχουν ε, ε, αλλάξει τελείως τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και κάποια παραδείγματα από το Πανεπιστήμιο του Λέστερ είναι στην ε, εγκληματολογία όπου έχουμε φοιτητές από πολύ επικίνδυνα μέρη του κόσμου που δεν υπάρχει σύνδεση πάντα ίντερνετ και εδώ έχουμε κάποιους ε, φοιτητέ στρατιωτικού που με τα διάφορα σκηνητέ συσκευέ στα iPads, τους έχουν δοθεί μάλιστα iPad. Εδώ έχουμε ένα άλλο παράδειγμα από την αρχαιολογία που χρησιμοποιείται το iPad έξω ε, στο, στην ανασκαφή για να συλλέξουν δεδομένα. Συλλογική τώρα είναι η πρωτοβουλία ISPOT που κανεί μπορεί να ανεβάσει στοιχεία από τη χλωρίδα και την πανίδα για να προωθήσει επιστημονικά ενδιαφέροντα του, γενικού, του ευρύτερου κοινού. Αλλά είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται αυτά τα άπειρα δημόσια στοιχεία για να, για να βελτιώσεις τις δικές σου, τις δικές σου γνώσεις. Τώρα, μάθηση σε συγκεκριμένες ε, ε, καταστάσεις και ε, ρόλοι. Εκεί οι φοιτητέ μπορούν να κινηθούν στο εικονικό εργαστήριο, να κάνουν ε, βόλτα, να διαβάσουν. Και ένα άλλο παράδειγμα του Google είναι η βήθηση, βήθηση στην μάθηση. Εγώ ήθελα λοιπόν να μάθω Ισπανικά και σήμερα το πρωί, ας πούμε, έβαλα κάποιες πληροφορίες ότι ο διευθυντής ε, της ενημέρωσης είναι στα, στα Ισπανικά, για παράδειγμα, και εδώ τι μπορεί να κάνεις. Αν ε, κλικάρεις τις λέξεις αυτές, μπορείς να αλλάζεις ανάμεσα στα Ισπανικά και τα Αγγλικά. Μπορείς δηλαδή να βυθιστείς τη γλώσσα. Τώρα, τεράστιος αριθμός ε, μαθητών που δεν μπορούν ή δεν έχουν πρόσβαση ή δεν, μπορούν, δεν έχουν χρήματα για να σπουδάσουν και γι' αυτό και η UNESCO προωθεί τους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους έχουμε εκατοντάδες ε, αρχεία παγκοσμίω. Η αξιολόγηση τους δείχνει όμως πως δεν χρησιμοποιούνται όσο θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από τους φοιτητές και από τους ε, καθηγητές και γι' αυτό και βλέπουμε πώς ο κόσμος ε, χρησιμοποιεί αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και έχουμε φτιάξει και κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Μπορεί κανείς να το κοιτάξει αυτό, να δει ποια είναι η στρατηγική του για τους ανοιχτούς πόρους ε, και ποια είναι η ποιότητα των στοιχείων που δίνει. Σε ένα επόμενο project, ε, το Power Up, κάνουμε την καταγραφή των ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων. Έχουμε καταγράψει εκθέσει για 11 χώρες και έχουμε κάνει 7 μελέτες σε βάθος. Αν το πάτε στο Google θα τα δείτε, είναι διαθέσιμα όλα αυτά τα στοιχεία. Κάτω-κάτω εδώ βλέπετε ένα βίντεο του YouTube για να μάθετε το διάφορα πράγματα για το σχεδιασμό της μάθησης. Έχουμε πολύ κόσμο. Και τέλος, θα έλεγα ότι έχουμε δει μια αναποδόμηση της εκπαίδευσης στους πόρους στους ε, δρόμους μάθησης, στη στήριξη και την διαπίστευση. Και βλέπουμε νέα μοντέλα ανάμεσα στις, δύο, στις ε, ε, τα τέσσερα αυτά στοιχεία, δηλαδή ανοιχτή πιστοποίηση. Έχουμε ένα σύστημα σφραγίδων από τους συναδέλφους και έχουμε και το ανοιχτό πανεπιστήμιο. Υπάρχει ένα διεθνές, διεθνής όμιλος που μπορεί να πάει κανείς και να, ένας φοιτητής και να πει θέλω εγώ να με πιστοποιήσει το τάδε πανεπιστήμιο στην Νότια Αφρική, ας πούμε. Και έπειτα θα πρέπει νομίζω να σκεφτούμε ε, τι σημαίνει αυτή η διάσπαση της ε, ε, παιδείας. Ποια είναι τα τμήματα που θέλουμε εμείς να στηρίξουμε στην επίσημη παιδεία και ποιος είναι ο ρόλος μας ως παραδοσιακά ιδρύματα Τι σημαίνει να υιοθετήσουμε πιο ανοιχτές προσεγγίσεις. Αν σας ενδιαφέρουν τα όσα συζητήσαμε, έχουμε ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Θα σας αφήσω κάποιο φυλάδι εδώ, αρχίζει του χρόνου. Και έχω ένα βιβλίο που μόλις έχει εκδοθεί φέτος, τα τελευταία μέρες μάλιστα, που σας δίνουν πολύ περισσότερες λεπτομέρειες για τα όσα σας ανέφερα εγώ σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που με ακούσατε. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Και περνούμε στη δεύτερη ενότητα τώρα. Και πριν ε, παραδώσω το συντονισμό και την Προεδρία στην κυρία Βάρπαρα Μόζερ Μέρσερ, θα ήθελα να σας ανακοινώσω απλώς ότι μας ρώτησαν ορισμένοι συμμετέχοντες εάν ε, θα υπάρχουν οι παρουσιάσεις ε, που ακούσαμε αυτό το διήμερο στην ιστοσελίδα μας. Έχουμε όλα τα στοιχεία. Έχουμε όλες τις παρεμβάσεις και θα παρακαλούσα όλους τους ομιλητές να μας πούν ότι αν κάποιος έχει αντίρρηση να ε, δημοσιευθούν οι παρουσιάσεις ε, στην ιστοσελίδα μας, να μας το δηλώσει. Υπάρχει δυνατότητα εξαίρεσης opt-out και σιωπή σημαίνει αποδοχή και συνένεση και θα είναι διαθέσιμα για όλους. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η Μπάρμπαρα Μόζε. Good morning and I know it's... Καλημέρα σας. Έχει ε, διαρκέσει ήδη πολύ το πρωινό. Παρ' όλα αυτά θα θέλαμε να κλείσουμε την πρωινή ενότητα πριν περάσουμε στα συμπεράσματα με κάποια παραδείγματα για το πώς χρησιμοποιούμε την τεχνολογία για να ενισχύσουμε τη μάθηση. Είχαμε μια εξαιρετική επισκόπηση όλων των εργαλείων που σήμερα διαθέτουμε, αλλά τελικά θα πρέπει να αναρωτηθείτε και εγώ πώς θα τα χρησιμοποιήσω όλα αυτά και πώς θα τα εσωματώσω στη δική μου λειτουργία και τι όφελος τελικά θα έχω από τη χρήση αυτών των εργαλείων. Μου ζήτησαν να συντονίσω τη συζήτηση αρχικά, αλλά μετά μου ζήτησαν να σας δώσω και ένα σύντομο παράδειγμα για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία σε ε, εξαιρετικές περιπτώσεις και ακραίες ανθρωπιστικές ε, καταστάσεις. Αν μου επιτρέπετε, σύντομα... Α, όχι. Πρώτα εσείς. Καλά. Α, επειδή έχει ε, προβληθεί στην οθόνη, εντάξει, θα αρχίσουμε πρώτα από την Κατερίνα Δάρα Λέπουρα, που θα σας μιλήσει για τις εικονικές τάξεις, οικονομικά μαθήματα και ζητώ συγγνώμη που παρενέβη. Καλημέρα σε όλους σας. Θα μιλήσω ελληνικά. Και ε, αν δεν καταλαβαίνετε ελληνικά, βάλτε τα ακουστικά σας για να μας φανούν κινέζικα. Κυρίες και κύριοι Πριτάνης, ε, κύριοι και κυρίες καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα σας παρουσιάσω σήμερα τα προγράμματα ηλεκτρονικής εκμάθησης και εικονικής διδασκαλίας της Γενικής Διευθυνσιός μου. Προς το παρόν έχουμε δύο προγράμματα. Τις τάξεις της εικονικής διδασκαλίας και το Speech Repository. Για το Speech Repository θα ήθελα μόνο να αναφερθώ επιγραμματικά, διότι το θέμα καλύφθηκε από την κυρία Επίτροπο. Θα σας πω απλώς ότι έγινε πρόσφατα μία έρευνα η οποία κατέδειξε ότι είναι πολύτιμο στην ε, εκμάθηση της διερμηνίας. Είναι πάρα πολύ προσφυλές και αγαπητό και στους καθηγητές και στους φοιτητές οι οποίοι το χρησιμοποιούν. Ξεκίνησε το 2007 στη Γενική Διεύθυνση ΣΚΙΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πολύ γρήγορα όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε με λόγους, ομιλίες, όπως επίσης και συναδέλφους διερμηνείς, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την αξιολόγηση της δυσκολίας των λόγων που μπαίνουν στο repository, το περίφημο grading. Μιλάμε λοιπόν σήμερα πάρα πολύ για εικονικές τάξεις διδασκαλίας, για εικονική πραγματικότητα. Εγώ όμως είμαι εδώ για να σας αποδείξω ότι είναι μια πραγματική πραγματικότητα. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπετε τη διεξαγωγή μιας τάξεως εικονικής διδασκαλίας. Βλέπετε εδώ τους διερμηνείς του Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι οποίοι εδώ είναι έτοιμοι να αξιολογήσουν τους φοιτητές. Εδώ βρίσκεται η Λισαβόνα, εδώ βρίσκεται η Γενέβη, εδώ βρίσκεται η Πράγα και εδώ οι Βρυξέλλες με τους διερμηνείς των τριών θεσμικών οργάνων. Πώς ακριβώς πραγματοποιείται. Έχουμε έναν διερμηνέα ο οποίος εκφωνεί έναν λόγο στην Λισαβόνα, ο οποίος μεταφράζεται προς τα πορτογαλικά στη Λισαβόνα, προς τα γερμανικά στη Γενέβη και προς τα τσέχικα στην Πράγα. Οι αξιολογητές της Βρυξέλλες κρίνουν την απόδοση των φοιτητών. Εδώ βλέπετε τον καθηγητή ο οποίος εκφωνεί το λόγο και εδώ τον φοιτητή ο οποίος είναι έτοιμος να τον μεταφράσει. Έχουμε δύο είδη ε, τάξεων εικονικής διδασκαλίας, της πολυμερής και της διμερής. Οι πολυμερείς μας δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε και ταυτόχρονη και επακολουθητική διερμηνία, η επακολουθητική περνάει μέσω από video conference, από τηλεδιάσκεψη, ενώ η ταυτόχρονη περνάει μέσα από το web streaming. Πολύ σωστά μια συνάδελφος με είχε πει στο παρελθόν, αισθάνομαι λίγο σαν να είμαι στη Eurovision. Όχι με την έννοια ότι εμείς είμαστε εδώ για να πούμε πόσους βαθμούς δίνουμε για τα τραγούδια στις διάφορες χώρες, αλλά είμαστε για να πούμε, για παράδειγμα, ότι συνδέομαστε με την Πράγα και τα σχόλια που έχουμε να κάνουμε στον Τσέχο φοιτητή είναι τα εξή και αμέσως μετά στη Λισαβόνα τα σχόλια που έχουμε να κάνουμε για τα πορτοκαλικά είναι το εξή. Και έτσι συνεχίζει η όλη διεξαγωγή της τάξεως. Βλέπετε εδώ κάτω-κάτω ήταν η πανηγυρική παρουσίαση των, ε, της εικονικής διδασκαλίας στις πολιτικές μας αρχές. Βλέπετε τον Αντιπρόεδρο κύριο Μαρτίνες και τον αρμόδιο τότε για θέματα πολυγλωσσίας Επίτροπο κύριο Ορμπάν και βεβαίως τους Γενικούς Διευθυντές. Πολυμερείς ε, τάξεις εικονικής διδασκαλίας διεξάγουμε με τα εξή πανεπιστήμια. Καταρχήν με τη Γενέβη, πανεπιστήμιο πρωτοπόρο στο χώρο της ηλεκτρονικής εκμάθησης και της εικονικής διδασκαλίας, τη Λισαβόνα, την Πράγα, την Εζίτ στο Παρίσι, τον Μπογκατζίση στην Τουρκία, τη Λουμπλιάνα και δύο καινούργια μέλη που είναι το Κλούς στην Ρουμανία και η Βουδαπέστη. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω αυτά τα δύο καινούργια μέλη στον κλαμπ των, ε, της εικονικής διδασκαλίας. Οι πολυμερείς τάξεις εικονικής διδασκαλίας απαιτούν φοβερή πειθαρχία, διότι καταλαβαίνετε ότι είμαστε συνδεδεμένοι με τρία διαφορετικά κράτη, με τρία διαφορετικά πανεπιστήμια, με φοιτητές οι οποίοι έχουν διαφορετικούς συνδυασμούς γλωσσών. Οπότε πρέπει όλοι να ακολουθούμε πολύ πιστά το σενάριο, το πρόγραμμα, το οποίο εκ των προτέρων έχει καταρτιστεί. Μάλιστα στη γλώσσα μας το, το αποκαλούμε script. Εγώ έχω την τάση το script να το γράφω μάλιστα με κεφαλαία για να τους δείξω ότι είναι η βίβλος που πρέπει με θρησκευτικό σεβασμό να ακολουθήσουμε. Βλέπετε, ας πούμε, για παράδειγμα, δεν φαίνεται καλά στη διαφάνεια, ότι για τις συστάσεις στην αρχή προβλέπουμε από τις 10 και 6 μέχρι τις 10 και 8 όχι ένα τέταρτο χοντρικά. Δηλαδή, είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ ακριβές. Και εδώ καθώς συνεχίζει βλέπετε ας πούμε ότι η διερμηνέας αρμόδια για να κρίνει τα τσέχικα έχει τον ίδιο συνδυασμό με τη φοιτήτρια η οποία βρίσκεται στην Πράγα. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί πολύ σωστά το σύστημα. Για οποιαδήποτε πληροφορία θέλετε για αυτού του είδους της τάξης σας παραπέμπω στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Γενέβης, η οποία αρχιοθετεί όλες τις τάξεις τις οποίες έχουμε πραγματοποιήσει μέχρι τώρα. Και βέβαια κάτι πολύ σημαντικό για αυτές τις πολυμερείς τάξεις είναι ότι εκτός από τους φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν ας την πούμε, στην πραγματική τάξη. Είναι και πάρα πολλοί άλλοι που συνδέονται μέσω web streaming και μπορούν να παρακολουθήσουν την τάξη. Μπορούν να υποφεληθούν από τους λόγους που εκφωνούνται από τους καθηγητές, όπως επίσης, ακόμα περισσότερο, από τις αξιολογήσεις που κάνουν οι διερμηνείς μας. Εδώ είναι πάντα η ιστοσελίδα της Γενέβης. Βλέπετε όπως πάντα την οθόνη χωρισμένη στα τέσσερα με την Γενέβη εδώ, τη Λισαβόνα και την Πράγα και εδώ ε, έναν πρώην συνάδελφό μου και εμένα είμαστε μάλλον στενοχωρημένοι και κατηφείς γιατί κάποιο τεχνικό πρόβλημα θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Δυστυχώς με την τεχνολογία τα απρόπτα υπάρχουν. Οι διμερείς τώρα ε, τάξεις ε, πρέπει να σα πω ότι είναι πολύ πιο οικίε, Αρέσουν πολύ περισσότερο στου φοιτητέ. Υπάρχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα συνέχεια, διότι ξέρουμε τον φοιτητή οπότε σε μια επόμενη τάξη μπορούμε καλύτερα να τον παρακολουθήσουμε. Ε, και βέβαια όταν δεν έχουμε να ακολουθήσουμε ένα τόσο αυστηρό σκρίπτ όπως έχουμε στις πολυμερείς ε, είναι όλα πιο εύκολα για όλους. Πραγματοποιούμε λοιπόν αυτού του τύπου τις τάξεις με το Κομίγια στη Μαδρίτη, με το Χέρτσεν στην Αγία Πετρούπολη, το Αστρακάν και το Φορλί στην Πολόνια. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα πανεπιστήμια τα οποία έχουν δυνατότητα να κάνουν διμερείς τάξης εικονικής διδασκαλίας, αυτή τη στιγμή εξετάζουμε το ενδεχόμενο πόσους περισσότερους θα μπορούμε να συμπεριλάβουμε στις τάξεις μας. Και βεβαίως υπάρχουν και πανεπιστήμια τα οποία έχουν ήδη αγοράσει τον εξοπλισμό και είναι έτοιμα από του χρόνου, για παράδειγμα έχω δύο πανεπιστήμια στην Πολωνία, τα οποία θα ήταν έτοιμα από του χρόνου να ξεκινήσουν και αυτά μαζί μας να κάνουν τις τάξεις εικονικής διδασκαλίας. Βέβαια, υπάρχει μία δυνατότητα, πολύ περιορισμένη, να κάνουμε και τάξεις μέσω Skype. Ε, κάνουμε με τη Σόφια, με τη Στοκχόλμη, με το Ταλίν, το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω, διότι μετά τις Skype κλάσεις αποφάσισε να περάσει στην video conference. Ε, και βέβαια για όσους ακούτε ότι κάνουμε Skype classes, παρακαλώ μην με πάρετε τηλέφωνο να μου πείτε ότι θέλω μία Skype class αύριο το μεσημέρι και αύριο το απόγευμα και αύριο το βράδυ και αύριο τα μεσάνυχτα, επειδή είναι εύκολη σύνδεση μέσω Skype, διότι υπάρχει ένα θέμα ποιότητας στην εικόνα και στον ήχο με το Skype και υπάρχει βέβαια και ένα θέμα ε, διαθεσιμότητας των διαρμηνέων. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι αν θέλετε να έχουμε ε, τάξεις εικονικής ε, διδασκαλίας θα ήταν πολύ καλύτερα να εξοπλιστείτε με εξοπλισμό για τηλεδιασκέψεις, video conference equipment, ε, διότι μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε πολύ καλύτερη ποιότητα στον ήχο και στην εικόνα. Μπορούμε να είμαστε πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Υπάρχει καλύτερη συνέργεια μεταξύ φοιτητών, καθηγητών και εικονικών αξιολογητών εκ μέρους μας και βέβαια μπορούμε όλοι να συγκεντρωθούμε καλύτερα στη δουλειά που κάνουμε. Πολλές φορές τα πανεπιστήμια έρχονται και με ρωτάνε «Μα τελικά πόσο στοιχίζει αυτός ο εξοπλισμός». Αυτός ο εξοπλισμός στοιχίζει 10 με 15.000 ευρώ, ευρώ. Ε, εξαρτάται από χώρα σε χώρα και εξαρτάται από τις δυνατότητες που έχει η κάθε τοπική αγορά. Ε, το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι αξίζει να τον αγοράσετε, διότι μας δίνει τη δυνατότητα να συνδεόμαστε και να έχουμε την ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τις τάξεις εικονικής διδασκαλίας. Πολλά τα ωφέλη, πραγματικά πολλά και για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και για τους φοιτητές. Ενδυναμώνουμε καταρχήν την επαφή που υπάρχει μεταξύ πανεπιστημίων και ευρωπαϊκών θεσμών υπάρχει πολύ καλή ανταλλαγή απόψεων μεταξύ καθηγητών και εικονικών αξιολογητών. Και βέβαια οι φοιτητέ θέλουν πάρα πολύ να ακούν τα σχόλια τα οποία κάνουν οι συναδελφοί μου. Μου έχει συμβεί περιστατικό που υπήρχε, ιδίω στι αρχέ που είχαμε τα τεχνολογικά προβλήματα, τα τεχνικά συγγνώμη προβλήματα, υπήρχε περιστατικό που διακόπη η σύνδεση περίπου για μια ώρα και ο φοιτητή περίμενε εκεί μετά από μία ώρα για να μπορέσει να κάνει τη διερμηνία του και εμεί να τον αξιολογήσουμε. Δηλαδή δεν θέλουν να χάσουν ούτε λεπτό από αυτή την ευκαιρία που τους προσφέρουμε. Οφέλει και για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, διότι έχουμε τη δυνατότητα να διαδώσουμε το μήνυμα για την καλή ποιότητα και τα υψηλά, τις υψηλές προδιαγραφές που έχουμε στη διερμηνία. Βεβαίως τίθεται και το οικονομικό όφελος, το οποίο μας επιτρέπει μέσω της, αυτής της σύνδεσης να είμαστε παρόντες σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου, σε ναι. με, πολύ, με πολύ μειωμένο το κόστος. Και βέβαια οι, ε, οι, οι, οι τάξεις διδασκαλίας έχονται και αυτές να συμπληρώσουν το πρόγραμμα το οποίο ισχύει ήδη εδώ και πολλά χρόνια της παιδαγωγικής στήριξης που πραγματοποιούμε. Θα τελειώσω με ένα όνειρο. Ε, ξέρετε ότι αν δεν έχουμε οράματα, εάν δεν είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις στο μέλλον, η τεχνολογία θα μας ξεπεράσει και μετά θα είναι πολύ δύσκολο να καλύψουμε το κοινό. Έλεγα λοιπόν ότι θα ήθελα ή δυνατόν να κάνουμε διάφορους συνδυασμούς κατά τη διάρκεια της δεξιαγωγής ε, της ε, εικονικής διδασκαλίας, εγώ, για παράδειγμα, είχα σκεφτεί μια ιδέα, θα ήταν να συνδέσουμε ένα πανεπιστήμιο EMCI στην Ευρώπη, ένα πανεπιστήμιο το οποίο δεν είναι EMCI, όπως για παράδειγμα το Φορλή στην Ευρώπη, και το Άστρακαρ ή το Πογκατζή στην Κωνσταντινούπολη. Η Γενική Διευθύντρια με ξεπέρασε, διότι ήρθε χτες και κατέθεσε μία πρόταση, προκειμένου να συνδεόμαστε με έναν ακόμα διεθνή οργανισμό και δύο πανεπιστήμια. Ε, πάρα πάρα πολύ καλή ιδέα. Ελπίζω μόνο να λάβουμε τουλάχιστον υπόψη μας τη διαφορά ώρας και να μην χρειαστεί να κοιμηθούμε στο virtual classroom προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις τάξεις εικονικής διδασκαλίας. Η δεύτερη μου επιθυμία θα ήταν να, να γίνουμε ακόμα τεχνικά καλύτεροι όσο αναφορά της, ε, όσον αφορά την ταυτόχρονη διερμηνία. Διότι εκεί είναι δυστυχώς που αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα ακόμα. Πολλές φορές η διερμηνία έρχεται με κάποια δευτερόλεπτα καθυστέρηση και έτσι δεν επιτρέπει στον εικονικό αξιολογητή να μπορέσει να ε, κάνει σωστή αξιολόγηση του φοιτητή. Και επειδή βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια των τεστ και των διαγωνισμών οι φοιτητέ κυρίω, οι υποψήφοι μάλλον σε αυτή την περίπτωση, δεν τα καταφέρνουν πολύ καλά με την ε, ταυτόχρονη διερμηνία, νομίζω ότι θα πρέπει αρκετά να επικεντρωθούμε και εκεί. Πριν τελειώσω και σας ευχαριστήσω, θα ήθελα πάρα πολύ να ευχαριστήσω τους τεχνικούς μας, της δικής μας Γενικής Διευθύνσεως, επίση και της DGITEC, για όλη τη βοήθεια που μας έχουν προσφέρει αυτά τα χρόνια προκειμένου να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε την εικονική διδασκαλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ θερμά, Κατερίνα. Πραγματικά ήταν πολύ πλήρης και εμπεριστατωμένη η επισκόπηση αυτών των δυνατοτήτων των τάξεων εικονικής διδασκαλίας, των πολυμερών, των διμερών. Εμείς τη λέμε και MVC είναι πολύ πιο εύκολο και πιο σύντομο με τα αρχικά. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στη Σουζάνε Άλτεμπεργκ για να μας δώσει το δικό της πρίσμα για το ίδιο θέμα. Ευχαριστώ πολύ Μπάρμπαρα. Πάρα πολύ σύντομα θα ήθελα να συμπληρώσω λίγο γιατί ξέρω ότι έχει να σας πει κάτι πολύ ενδιαφέρον να μας πει η Μπάρμπαρα Μόζε. Γι' αυτό ε, από εκεί που σταμάτησε η Κατερίνα θα ήθελα λίγο να συμπληρώσω μερικά πράγματα γιατί έχει σημασία να πούμε ίσως ότι θέλουμε να επεκτείνουμε ακόμα περισσότερο την ηλεκτρονική εκμάθηση, το e-learning είναι ε, ένα κέντρο βάρους, γι' αυτό υπάρχει και ένα νέο τμήμα και θέλουμε να ενισχύσουμε στη Γενική Διεύθυνση την όλη αυτή διαδικασία. Και πέρα από τις εικονικές ε, τάξεις, δεν ξέρω και πώς θα το λέγαμε στα γερμανικά, ε, εικονικές ε, τάξεις, λοιπόν, masterclass, θέλουμε να έχουμε και ένα είδος εικονικής ε, παρακολούθησης, coaching για εκείνους που σπουδάζουν, που ε, έχουν δυναμικό και που μας ενδιαφέρουν λόγω του γλωσσικού συνδυασμού τους για εργασία. Και αυτό μπορεί να γίνεται και ταυτόχρονα και με χρονική στέριξη ηλεκτρονικά. Θα πρέπει να τα δούμε όλα αυτά ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. Βεβαίως υπάρχει επικουρικότητα στην εκπαίδευση, τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για θέματα παιδείας, αλλά εμείς επιθυμούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και εργοδοτών. Αυτό υπάρχει ήδη στην ιδιωτική οικονομία, αλλά στους δημόσιους θεσμούς ίσως δεν έχει προχωρήσει, δεν είναι τόσο διαδεδομένο. Γι' αυτό θα θέλαμε και με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών και της ηλεκτρονικής διδασκαλίας και να εξασφαλίσουμε τη μετάβαση από τις σπουδέ στην εργασία. Η Κατερίνα αναφέρθηκε στις τεχνικές προϋποθέσεις, δεν είναι και τόσο φθηνό. Θα ήθελα να σας πω ότι στα πλαίσια του προγράμματος επιδοτήσεων για τα προγράμματα των πανεπιστημίων, το διαθεσμικό υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης και η χρήση νέων τεχνολογιών είναι και σημαντικό κριτήριο. Γι' αυτό θα ήταν ε, και αυτή μια δυνατότητα υποστήριξης οικονομικής. Πέρα από τη φάση της εκπαίδευσης στο ίδιο το Πανεπιστήμιο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για ε, τα τεστ ε, επιλογής ε, υποψηφίων διερμηνέων και προεπιλογής ήδη για τέτοια τεστ κατά τα κτίρια έχουμε κάνει εξαποστάσεως. Ε, τέτοια τεστ ή ακόμα όταν κάποιος δίνει για να πάρει υποτροφία να μάθει μια γλώσσα. Ε, αυτά ήθελα να πω εγώ. Ένα σημαντικό στοιχείο για κάθε είδους e-learning είναι ότι αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο οι οικονομίες, ε, η υπόθεση του περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, μειώνονται τα ταξίδια, ε, μειώνεται το αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα, είναι φιλική στο περιβάλλον και στις μελλοντικές γενιές αυτή η μορφή εκπαίδευσης και θα μπορέσουν να ε, συνηθίσουν και οι νέες γενιές διερμηνέων στις νέες τεχνολογίες. Γιατί μετά από όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα, και τελειώνω αυτό, θα ήθελα να πω τύπο Bill Good ότι είναι γεγονός ότι δεν θα αντικατασταθούν ή δεν θα αντικατασταθούν αύριο οι διερμηνείς από τεχνολογία αλλά από άλλους διερμηνείς που χρησιμοποιούν την τεχνολογία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Σουζάνα για τι εμπληρώσεις αυτές ε, στην παρουσίαση της Κατερίνα. Μας έδωσες και μια πρόπτικη για το μέλλον. Επιστρέφω στα αγγλικά τώρα. Απλώς για να σας δείξω ότι μιλάω και γερμανικά ήταν αυτό. Θα ήθελα να δώσω όλη συνέχεια στις δύο παρουσιάσεις που ακούσαμε μόλις τώρα, καθώς και τις πρωινές, για να σας μεταφέρω σε ένα άλλο κόσμο. Μας πήγε η καθηγητής Βάιμπλ κάπου σε αυτό το προορισμό σήμερα το πρωί και θα αναφερθώ και στα λεγόμενά του. Επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω κάπου αλλού, σε ένα άλλο ταξίδι που πολύ συχνά κάνω αυτές τις μέρες. Έχω βγει από το ενιδρίο, αλλά όχι για πάντα, επιστρέφω από καιρούς καιρό, αλλά ταξιδεύω και σε άλλα μέρη του κόσμου που χρησιμοποιείται διερμηνία και όπου η ποιότητα της διερμηνίας συνήθως δεν είναι πάρα πολύ καλή. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία για την επιβίωση ε, και τη μοίρα πολλών ανθρώπων είναι ζωτική σημασία. Θα ήθελα εδώ να το συνδέσω με διάφορα που ακούσατε σήμερα το πρωί. Η δυνατότητα χρήσης τεχνολογίας για να υπάρχει δυνατότητα ε, ανθρώπων να επικοινωνούν μεταξύ τους σε κατεπίγουσες καταστάσεις με τρόπο περιορισμένο αλλά πάρα πολύ σημαντικό. Ζωτική σημασία ε, για αυτό το θέμα της επιλογής ε, που ακούσαμε προηγουμένως που, ε, για να ξέρουμε πού θα στείλουμε τον κάθε ε, άνθρωπο και δεν μπορούν όλοι οι διερμηνείς να έρχονται σε επαφή με όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ χαότης γενικά γιατί είναι εκτακτή και επίγουσα. Στη συνέχεια θα ήθελα να το συνδέσω και με αυτό που ακούσαμε από τον Αλέξη σήμερα το πρωί για το πώς χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες εκμάθησης για την απόκτηση δεξιοτήτων. Γιατί σε τελική ανάλυση οι διερμηνείς χρειάζονται δεξιότητες και είδαμε πώς αλλάζει ο εγκέφαλος, πώς μαθαίνει να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Οπότε, ό,τι ξέρουμε για τον τρόπο εκμάθησης των δεξιοτήτων τελικά θα πρέπει να μεταφραστεί και στη λήψη των αποφάσεων που πρέπει να πάρουμε εμείς ως εκπαιδευτές. Δηλαδή, ποια είναι εκείνα τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε. Η καθηγήτρια Κονέλ μας παρουσίασε μια σειρά εργαλείων που υπάρχουν και πολλά από αυτά υπάρχουν, πώς να το πω, σε περιβάλλοντα που βρίθουν ε, τεχνολογίες. Ε, έχουμε ε, πολλές επιλογές, μεγάλη δυνατότητα διασύνδεσης παντού στο διαδίκτυο και στο τηλέφωνο να πιάνει 5 στα 5 όπου και να πάει κανείς, αλλά δεν είναι πάντα αυτή η χώρη που γίνεται η διδασκαλία και μάλιστα ηλεκτρονική διδασκαλία και εικονική. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα εγώ να σας δείξω είναι πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις νέες τεχνολογίες ως μοχλό και σε ακραίες περιπτώσεις και συνθήκες και ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις να έχετε όφελος από τις τεχνολογίες. Δεν θα επικεντρωθώ πάρα πολύ στο δικό μας έργο, ε, στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης γενικά, αλλά ε, συγκεκριμένα θα ήθελα να αναφερθώ ε, στην εικονική εκμάθηση. Δεν ξέρω αν είχα την ευκαιρία να το συζητήσω μαζί σας. Υπάρχει μια απόχρωση που θα μπορούσαμε, θέλετε, να συζητήσουμε κατά τη διάρκεια ε, του διαλύματος για καφέ, αν έχουμε και άλλο τέτοιο διάλειμμα. Λοιπόν, πώς ε, βρίσκουν εφαρμογή τεχνολογίες στην εκπαίδευση για την υποστήριξη των ε, μαθητών και των φοιτητών και πώς εγγράφεται η τεχνολογία στην υπηρεσία της παιδαγωγικής. Γιατί εγώ από αυτό τον κλάδο προέρχομαι, είμαι εκπαιδευτικός και με το νέο αυτό πρόγραμμα που έχουμε Έχω πάρα πολύ λίγο χρόνο για να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, πώς τα καταφέρνουμε όλα αυτά. Ε, μία παράθεση, έχω πολλές. Η έλλειψη μετάφρασης και διερμηνίας είναι ο βασικός ελίπων ε, κρίκος στη δυνατότητά μας να ε, συντονίζουμε ανθρωπιστική βοήθεια με τρόπο αποτελεσματικό και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο βελτίωσης της κατάστασης αυτής. Όπως θα γνωρίζετε στις ανθρωπιστικές ε, καταστάσεις, πολλές μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλοι οργανισμοί χρειάζονται συντονισμό στην παροχή βοήθειας. Είναι πάρα πολύ ακριβώς αυτός ο συντονισμός και κοστίζει και ζωές, γιατί όσο περισσότερο διαρκεί η διαδικασία λήψη αποφάσεων, τόσο περισσότερος κόσμος πεθαίνει. Ένας από τους βασικούς φραγμούς είναι ο γλωσσικός φραγμός για την έλλειψη συντονισμού. Εάν δεν μπορείς να συνεννοηθείς, να μιλήσεις με μια οργάνωση που λειτουργεί δίπλα σου, προφανώς δεν μπορεί να συντονιστείς. Και εκεί κοστίζει ζωές η γλώσσα ίδια. Ε, τόσο δεινή είναι η κατάσταση και τόσο εκτρή. Χρειάζεται λοιπόν σε περίπτωση θεομηνιών μεγάλο συντονισμό και θεομηνίες μπορεί να είναι είτε φυσικές καταστροφές είτε ε, ένοπλες Αναπτύσσουμε λοιπόν το έργο αυτό στο τμήμα διερμηνίας και κοιτάξαμε την κατάσταση από τρεις διαφορετικές αφετηρίες. Είπαμε ότι θέλουμε να γνωρίζουμε περισσότερο για το τι συμβαίνει πραγματικά επί τόπου και οι διερμηνείς, ο κλάδος, επάγγελμα αφιέρωσε πολύ χρόνο στη συλλογή στοιχείων. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος για να φτάσουμε στους εκπαιδευτές. Δεν είναι συνάδελφοι που μπορούμε να φέρουμε στη Γενέβη, στις Βρυξέλλες ή δεν ξέρω σε κάποια άλλη πόλη και να τους εκπαιδεύσουμε. Άρα θα πρέπει να πάμε εμείς εκεί. Είτε οι ίδιοι, είτε εικονικά ή με κάποιον άλλο τρόπο. Και τρίτον, μάθαμε ότι οι διερμηνείς που εκπαιδεύτηκαν, ας πούμε, στο Ουσμπεκιστάν ή άλλοι που εργάζονται στο Σοδάν ή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, φαίνεται ότι έχουν πολλά κοινά, οι ανάγκες τους δεν είναι ουσιαστικά πολύ διαφορετικές. Άρα ε, πώς θα τους φέρουμε σε επαφή. Μπορούμε να δημιουργήσουμε εικονικές ε, επαγγελματικές ε, κοινότητες. Ίσως να σας κάνει εντύπωση που χρησιμοποιώ τον όρο επαγγελματίας για μη εκπαιδευμένους διερμηνείς. Συνειδητά το χρησιμοποιώ και θα σας πω και σε πόσες γλώσσες συμβαίνει σε λίγο. Και αν έχω χρόνο, θα αναφερθώ σε αυτό το ζήτημα που είναι όντως ε, λεπτό και ευαίσθητο. Λοιπόν, αυτό είναι το έργο μας, το πρόγραμμα που εκπονήσαμε και τι κάνουμε. Εντοπίζουμε τις ανάγκες των διερμηνέων που εργάζονται σε ζώνες εμπόλεμες και, και τις δικές μας ανάγκες. Ε, σχεδιάζουμε ε, τρόπο εκπαίδευσης, τους εκπαιδεύουμε εικονικά ε, αλλά και με κάποια προγράμματα προσχεδιασμένα. Το έχουμε κάνει με τον ε, Ερυθρό Σταυρό αυτό. Τους τελευταίους 12 μήνες έχω πάει πολλές φορές επί να αρχίσω την εκπαίδευση και μετά συνεχίζουμε με τρόπο εικονικό όταν φεύγουμε. Αξιολογούμε και τα μαθήματα και τις ε, ικανότητες και κάνουμε εταιρικέ σχέσεις με τα τοπικά πανεπιστήμια, γιατί δεν είναι μόνο η ανθρωπιστική διάσταση, υπάρχει και η αναπτυξιακή διάσταση. Και ανάπτυξη σημαίνει οτιδήποτε ε, αρχίζει από βορρά προς νότο, κάποια στιγμή θα πρέπει να έχει φορά από το νότο προς τον νότο. Ε, γιατί φαίνονται και συμφέρουν οι επιχείρησεις αυτές, έχουν συμφέρον μάλλον τα πανεπιστήμια να συνεργάζονται μεταξύ τους. Ας πούμε, το Ναϊρόμπι, το πανεπιστήμιο με το πανεπιστήμιο της Χαρτούμ. Και ε, του φέρνουμε σε επαφή για να ε, προωθηθεί αυτή η συνεργασία. Όταν βγαίνεις λοιπόν από το ενιδρίο, αλλάζει λίγο η κατάσταση. Θα έχετε δει ε, αυτά τα ονόματα που σας δείχνω και στον τύπο. Και εδώ προσπαθώ να σας εξηγήσω πώς λειτουργούν αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Ανάλυση πρώτα των αναγκών. Τώρα έχω μπει ήδη στο περιεχόμενο, στην ουσία. Ανάλυση των αναγκών λοιπόν. Στην τριετία που εργαζόμαστε σε αυτό με πιο εντατικούς ρυθμούς, οι ανάγκες ε, γενικά εντάσσονται σε δύο κατηγορίες. Το ένα είναι να υπάρχουν δεξιότητες διερμηνίας στην επακολουθητική διερμηνία και το άλλο είναι η δεοντολογία. Ποιος είμαι, τι ρόλο παίζω, τι χρειάζεται ο κόσμος από μένα και τι θα πρέπει να κάνω και κυρίως τι δεν πρέπει να κάνω. Αυτά ε, είναι τα δύο μαθήματα που έχουμε επεξεργαστεί. Εδώ είναι η επαγγελματική διοντολογία. Ε, περιγραφή του μαθήματος. Δείχνει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο που προσπαθούμε να διδάξουμε και κάθε μάθημα μετά κατανέμεται, κάθε διδακτική μονάδα αν θέλετε, σε πολύ διαφορετικές ε, διδακτικές δραστηριότητες. Εδώ στη δεοντολογία ε, λέμε ρητά τους στόχους μας, το περιεχόμενο που καλύπτουμε, το πρόγραμμα ε, για τη συγκεκριμένη κοινότητα, πώς αξιολογούμε τις ικανότητες και δεξιότητες και ποιοι είναι οι καθηγητές. Εδώ πρόκειται για το Χαρτούμ και το Ανατολικό Σουδάν. Πριν από δύο εβδομάδες ε, είχαμε ένα πρόγραμμα δεκαετούς εκπαίδευσης διερμηνέων που εργάζονται και στο Χαρτούμ και στις διάφορους προσφυγικούς καταβλισμούς στα σύνορα του Σουδάν και την Ανατολική περιοχή. Στον Ταρφούρ δεν πήγαμε για λόγους ε, ασφαλείας. Το Ανατολικό Σουδάν είναι λιγότερο επικίνδυνο κάπως και ε, μας έδωσαν την άδεια να μεταβούμε εκεί. Αλλά για να σας δώσω μια ιδέα για το πώς εργαζόμαστε εκεί. Όταν πήγαμε και ε, στήσαμε όλο το πρόγραμμα, μας είπαν ότι η Σουδανική κυβέρνηση ε, έβαλε ένα νέο κανόνα ότι χρειαζόσουν οπωσδήποτε άδεια για να πάει στην ε, ανατολική περιοχή της χώρας, πέρα από τη θεώρηση διαβατήριων που χρειάστηκε έτσι και αλλιώς χρόνο και κόπο για να τη πάρουμε. Και δύο μέρες περιμέναμε σε ένα ξενοδοχείο και αυτό συνέπεσε με τις διαδηλώσεις μετά τη δημοσίευση των ε, γελιογραφιών και είπα τη αρμοστία για τους πρόσφυγες για την οποία εργαζόμουν μας κράτησε εκεί στο ξενοδοχείο. Τελικά διαμαγείας ήρθε η έγκριση και η άδεια και όλοι εξεπλάγησαν. Και μάλλον επειδή είμαστε από πανεπιστήμιο και η παιδεία ε, φαίνεται ε, είναι ακόμα αρκετά ουδέτερη. Ε, δεν θα πρέπει να ξεχνούμε το είδος της επιρροής που έχουμε εμείς πανεπιστημιακοί και γενικά τα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε τέτοιες καταστάσεις. Ε, λοιπόν, όπως σας είπα, έχουμε τις διάφορες ε, δραστηριότητες, εκμάθησης, αναλύουμε ποια είναι τα σενάρια διερμηνίας. Αν κανείς έχει πάρα πολύ λίγο χρόνο να εκπαιδεύσει έναν υποψήφιο πρέπει να ξέρει ακριβώς τι θα κάνει. Δεν έχεις μήνες, έχεις δύο μέρες. Οπότε κάθε δραστηριότητα θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σαφώς περιγεγραμμένη. Ε, τους ίδιους στόχους έχουμε για τις ίδιες ασκήσεις. Αλλά αν δώσω την ίδια άσκηση σε κάποιον από την ύπατη ε, αρμοστία είναι πως κάνεις τη συνέντευξη για να δεις αν είναι κάποιος πρόσφυγας. Ενώ πηγαίνοντας στην Καμπούλ ε, μπορεί να είναι η συλλογή στοιχείων για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο στόχος δεν αλλάζει, αλλάζει το περιεχόμενο και ο τρόπος με τον οποίο εργαζόμαστε είναι ο ίδιος. Για να βεβαιωθούμε ότι ο διερμηνέας είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος για τη συγκεκριμένη δουλειά και ό,τι του προσφέρουμε έχει νόημα για τον ίδιο. Άρα πρέπει να είναι πολύ συγκεκριμένο το περιεχόμενο. Δεν θα επεκταθώ πολύ περισσότερο. Ε, μερικά παραδείγματα μόνο να σας δείξω. Για το πώς επικοινωνούμε με τους ανθρώπους αυτούς. Η ε, καθηγήτρια Κονέλη είπε ε, το, το τηλέφωνο, ιδίως στην Αφρική, ε, είναι κάτι που, που πιάνει παντού. Πέντε στα πέντε στο, ε, το σήμα. Στο Σουδάν μπορεί να μην βρείτε στο σελίδα ή μπορείτε ε, να μπείτε πιο εύκολα στην Κένια. Ε, και όλα αυτά θα πρέπει να τα λαμβάνετε υπόψη στην εκπαίδευση. Αυτές οι μικρές λεπτομέρειες έχουν σημασία. Επίσης μπορεί να διαπιστώσετε ότι για τη διεθνή κοινότητα τον, του Ερυθρού Σταυρού οι διερμηνείς είναι υπάλληλοι, ενώ σε θέματα προσφύγων ε, είναι πολλές φορές ντόπιοι ε, και υπάρχουν θέματα ασφαλείας, ας πούμε μπορεί, χρειάζεται να δανείζονται άλλο όνομα ή ε, να είναι ανώνυμοι και παρόλα αυτά να τους εκπαιδεύετε. Επίσης να μην δείχνετε φωτογραφίες τους. Υπάρχουν μια σειρά θεμάτων που πρέπει να λαμβάνετε υπόψη και αυτός είναι ο κατάλογος των μαθημάτων που κάνουμε. Και για κάθε δραστηριότητα, για κάθε δράση, έχουμε φόρουμ ε, με ανταλλαγή. Είναι χαμηλής τεχνολογίας, αλλά παρόλα αυτά έχουν πρόσβαση διερμηνείς και βλέπετε εδώ πώς επικοινωνούν, αλλάζουν, ανταλλάσσουν απόψεις και πώς έρχεται ο καθηγητής από τη Γενέβη και τους απαντάει με feedback, με αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της δραστηριότητας ε, που συμμετέχουν. Βλέπετε, ο συμμετέχων είναι ανώνυμος, ο καθηγητής είναι επώνυμος. Τώρα προσπαθούμε να αναπτύξουμε κάποιες κοινότητες και κάποιες πρακτικές και όπου έχουμε αρχίσει ε, στα πλαίσια της είπα της αρμοστίας για τους πρόσφυγες ε, μπορούν να ε, επικοινωνούν μεταξύ τους στο αϊρόμπι, Χαρτούμ, ε, καταβολισμοί, προσφύγων ε, στα πλαίσια της ΥΠΑ της Αρμοστίας εντός της ίδιας οργάνωσης. Ακόμα υπάρχουν φραγμοί μεταξύ των διαφόρων οργανισμών για λόγους προφανείς που δεν θέλω να σας αναφέρω σε λεπτομέρειες. Μπορείτε λοιπόν να δείτε ότι στη Γενέβη έχουμε πολλά περιβάλλοντα ας διδασκαλίας και εκμάθησης. Ε, εδώ δεν θέλουμε να έχουμε μεγάλη τεχνολογία, μεγάλα αρχεία, ε, που να χρειάζεται να κατεβάζουν και να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ε, ε, τους δίνουμε CD που δεν χρειάζεται να τυπώσουν μετά. Στέλνουμε από την Γενέβη τα σχόλια μας στους καταφλισμούς και ε, στη Βόρεια Κένια αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολύ ενθουσιώδης. Ε, έναν υπολογιστή έχουν και στον έναν υπολογιστή ε, κάνει ο καθένας τη δουλειά του και πραγματικά αυτά τα προβλήματα που έχουμε δεν θα πρέπει να γίνονται εμπόδια. Κάθε φορά θα πρέπει κανείς να μελετάει την ιδιαιτερότητα της κατάστασης και η παιδαγωγική προσέγγιση του να είναι αντίστοιχη με το πλαίσιο που καλείται να λειτουργήσει. Ας πούμε, ξέρουμε τι κάνουμε για την απόκτηση δεξιοτήτων και μπορούμε μέσα σε λίγες μέρες να διδάξουμε αυτό που θέλουμε. Μπορεί η Κλοντιρό να θέλει μια φωτογραφία που έφερα μαζί μου πρόσφατα. σας δείξω πώς γίνεται η λήψη των σημειώσεων για την επακολουθητική διερμηνία. Χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα ως φωτογραφική μηχανή. Παίρνουν φωτογραφίες δηλαδή από τις σημειώσεις και μετά εμείς τους στέλνουμε οδηγίες από τη Γενέβη. Ε, στην αρχή σημειώνω ακόμα πολλά λέξεις, και μετά στο τέλος έχουμε ένα παράδειγμα μια ομιλίας 2,5 λεπτών που πήρε σημειώσει ένα συμμετέχων στην Χαρτούμ πριν από λίγες εβδομάδες. Μία μάλλον ε, διερμηνέας που είναι αραβόφωνη ε, και ε, γράφει από δεξιά προς τα αριστερά όπως βλέπετε. Ήταν η ιστορία ενός πρόσφυγα πώς έγινε μια επίθεση ένα πρωί, πώς ε, ο κόσμος κυκλοφορούσε στους δρόμους, φώναζε, βλέπετε τις εικόνες. Χρησιμοποίησαμε αυτά τα στοιχεία και με δικού μας φοιτητέ στη Γενέβη για να τους δείξουμε ότι μπορεί να υπάρχουν πολιτιστικέ διαφορές αλλά οι σημειώσει για την επακολουθητική πολλές φορές ε, ε, δεν έχουν σχέση με τη γλώσσα και ήταν πάρα πολύ καλή και η διερμηνία της συγκεκριμένης φοιτήτριας. Επίσης βοηθούμε και άλλες οργανώσεις, όπως αυτή την περίπτωση είναι κέντρο τεχνολογικό του Ιδρύματος Δον Μπόσκο και μπορούν να πάνε εκεί οι δερμηνείς μας και να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις. Ήθελα να σας δείξω και αυτό, αυτή τη φωτογραφία γιατί αναφέρθηκε το θέμα των συναισθημάτων έχουμε βρει και γι' αυτό παιδαγωγικές ε, προσεγγίσεις ε, και εξ αποστάσεως και επιτόπου, αλλά δεν θα επεκταθώ. Εδώ ζουν οι δερμηνείς Για να έχετε μια ιδέα και τις διαμονής. Προσπαθούμε να βρούμε ένα μπούσουλα για το μέλλον. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι ότι μπορούμε με την τεχνολογία που δίνουμε να κάνουμε τη διαφορά και να βοηθήσουμε αυτούς τους συμμετέχοντες. Πάνω από 100 είναι τώρα στο διαδίκτυο online και πολλοί ενδιαφέρονται να πάρουν και ένα πιστοποιητικό ε, ανθρωπιστικής διερμηνίας που ε, αυτή τη στιγμή εκπονούμε και ελπίζουμε να ολοκληρώσουμε και του χρόνου να ε, βγει και στο διαδίκτυο. Εικονικό θα είναι, ελπίζουμε να αναβαθμίσει την επαγγελματική στάση και τα προσόντα των διερμηνέων που εργάζονται και ευχαριστώ. I think the uh, Ευχαριστώ. Μια και είμαι και συντονίστρια, κρατάω το προνόμιο του μικροφόνου. Δεν ξέρω αν μας έχει περισσέψει λίγος χρόνος για ερωτήσεις. Ναι, αλλά για πολύ σύντομες. Τρεις μόνο παρακαλώ και λακωνικές. Ο Χάρη από το Κινέζικο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών. Έχω μια ερώτηση προς την Κατερίνα και θα την κάνω στα Κινέζικα. Μιλήσατε για την επιθυμία σας να διευρύνετε τη συμμετοχή σε αυτές τις τάξεις εικονικής ε, διδασκαλίας. Μία ερώτηση λοιπόν. Θα συμπεριλάβετε και πανεπιστήμια εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κινέζικο Πανεπιστήμιο για παράδειγμα, όπω το δικό μας. Και αν η απάντησή σας είναι καταφατική, πείτε μας κάποιες λεπτομέρειες. Τι προϋποθέσεις ε, χρειάζονται, ε, ποιο είναι ένα σημείο επαφής, κάποια στοιχεία που θα μπορέσετε να μας δώσετε, κάποιες λεπτομέρειες. Ε, Σουζάν, είμαστε κι εμείς επιλέξιμοι για χρηματοδότηση τέτοιων πρωτοβουλειών. Φαντάζομαι ότι σε τέτοια περίπτωση θα ήμασταν πολύ ευχαρίστως να αγοράσουμε τέτοιου είδους ε, προϊόντα ευρωπαϊκά. Ευχαριστώ, Χάρη, πάρα πολύ σύντομα να απαντήσω. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορείτε να τα συζητήσετε διμερώς με την Κατερίνα και σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση φοβάμαι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή δυνατότητα γιατί ε, προς το παρόν περιορίζεται αυτό στις χώρες της Ένωσης και τις υποψήφιες προς ένταξη. Αλλά θα το έχουμε υπόψη μας και θα ε, είπα ότι εξετάζουμε το ενδεχόμενο να διευρύνουμε τον κύκλο των πανεπιστήμιων με τα οποία συνεργαζόμαστε και διευκρίνησα ότι υπάρχει και ένα πρόβλημα διερμηνέων. Πρέπει να δούμε αν υπάρχουν διερμηνείς διαθέσιμοι για να μπορέσουν να προβούν στην αξιολόγηση των γλωσσών των φοιτητών σας. Ε, αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε διμερώς και να, να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Σουζάννα Έρη και Νοέλ Μόιλε. Η Σουζάννα πρώτα. Ευχαριστώ. Με την άδειά σας θα μιλήσω ισπανικά. Συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του πάνελ. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσε οι παρουσιάσει. Έχω μια σύντομη ερώτηση προ την Μπάρμπαρα. Για ποιο λόγο αποφασίσατε να περάσετε από, το, από την απόλυτα ηλεκτρονική εκμάθηση στις ε, προσωπικές ε, εκπαιδευτικές ε, συνεδρίες και μετά να χρησιμοποιήσετε την ηλεκτρονική εκμάθηση. Ποιος ο λόγος μετάβασης. Κάναμε ε, λεπτομεριακή αξιολόγηση του αμυγός εικονικού μοντέλου και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το πλαίσιο στη, της διερμηνίας, της ανθρωπιστικές τέτοιες επιχειρήσεις ήταν πολύ περίπλοκο και δεν μπορούσαμε να καλυφθούμε μόνο από εικονικές ε, μεθόδους ε, διδασκαλίας γιατί έχουμε και τα διάφορα συναισθηματικά ε, τραύματα, την κόποση της συμπόνιας, όλα αυτά επηρεάζουν το έργο των διερμηνέων Γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε το συνδυασμένο μεικτό μοντέλο. Άλλωστε δεν επιμορφώνουμε μόνο διερμηνείς, γιατί δεν αρκεί κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε και τους χρήστες. Και είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τους τελευταίους 8 μήνες, όπου και αν πήγαμε, είχαμε 100% των χρηστών ε, παρόντες στο σεμινάριο γιατί ενδιαφέρονται και οι χρήστες για τη διερμηνία. Ε, συζητούμε κυρίως τα διοντολογικά θέματα μαζί τους. Και όλα αυτά, <laughs> την πολιτή μου πείρα στο ενιδρίο, ανέκαθεν να είχα την επιθυμία να έχουμε τόσο ε, προσεκτικούς χρήστες που να λαμβάνουν τόσο πολύ υπόψη και τις δικές μας ανάγκες όπως το είδαμε στις ανθρωπιστικές ε, ενισχύσεις και τέτοιου είδους φυσικά πρωτοβουλίες δεν μπορούν να γίνουν μόνο εικονικά μέσω του διαδικτύου. Ο Νοέλ. Ευχαριστώ, Μπάρμπαρα. Εγώ δεν είμαι διερμηνέας, αλλά θα ήθελα να γίνω. Και μάλιστα προετοιμάζομαι, διαβάζω ε, βιβλία για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, για τους άλλους διεθνείς οργανισμούς και ή βρήκα και το speech repository, αυτό το αρχείο των ομιλιών. Θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω, δεν ε, ε, φοιτώ σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά για να έχω μια εμπειρία και να δω αν με εξυπηρετεί, θα ήθελα να το χρησιμοποιήσω. Μια απλή λοιπόν και πρακτική ερώτηση. Μπορώ να το κάνω, να χρησιμοποιήσω το speech repository. Υπάρχει μια steering committee, υπάρχει μια steering committee η οποία αποφασίζει την οποιαδήποτε εξέλιξη ε, θα ακολουθήσουμε στο Speech Repository και είναι πάρα πολύ σαφείς οι χρήστες, περιγράφονται πολύ σαφώς οι χρήστες του Speech Repository και ποιος έχει δυνατότητα πρόσβασης. Ε, δυστυχώς η κατηγορία που μου αναφέρεις δεν έχει δυνατότητα πρόσβασης. I think this is an issue και εμείς στο EMCI αντιμετωπίσαμε τέτοιες απορίες και το θέμα της πρόσβασης σε ε, τράπεζες ομιλιών, αρχεία ομιλιών και την πρόσβαση σε αυτές. Εδώ και καιρό το εξετάζουμε, αλλά ακόμη δεν έχουμε βρει λύση, γιατί είναι αρκετά περίπλοκο το πρόβλημα. Δεν είναι ότι είμαστε απρόθυμοι να ανοίξουμε την πρόσβαση, υπάρχει και θέμα πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ιδιαίτερα για τράπεζες ομιλιών που έχουν συστήσει πανεπιστήμια. Δεν θέλουν ε, οι εκπαιδευτές να κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο οι ομιλίες τους. Υπάρχουν θέματα copyright. Όλους αυτούς τους περιορισμούς θα πρέπει να τους λάβουμε υπόψη. Πάντως έχουμε αντιμετωπίσει και εμείς παρόμοια θέματα. Πριν περάσουμε στα τελικά σχόλια, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον καθηγητή Αράις. Αγαπητή κυρία Κοσμίδο θα ήθελα εκ μέρου του καθηγητού Σαλήμ Ντακάς, του Πριτάνος του Πανεπιστημίου του Αγίου Ιωσήφ στη Βηρητό, να σας δώσω το μετάλλιο του Πανεπιστημίου. Δυστυχώς ο καθηγητής αποσιάζει για προσωπικούς λόγους προσωπικού πέθους. Και για να σας κάνω την παρουσίαση θα ήθελα παρακαλώ να την κάνω στα αραβικά, γι' αυτό σας θέλω παρακαλώ να βάλετε τα ακουστικά σας. Κυρία Κοσμίδου, ε, αναζητάτε τερμινείς ε, όπως κάποιοι ε, αναζητούν σπάνια όστρακα στις αμμουδιές Στι ε, στις διάφορες παραλίες και ε, ψάχνετε τον καλό διερμηνή όπως κάποιος ψάχνει το σπάνιο αστρίδι με το μαργαριτάρι. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήρθατε στη Βηρητό να επισκεφτείτε τη σχολή μετάφραση και διερμηνίας. Είχατε επαφές με την ε, σχολή μας. Σας ευχαριστούμε θερμά και θα ήθελα να σας ε, εκφράσουμε την αναγνώριση και την ευγνωμοσύνη μας. Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, φτάσαμε αισίως στο πέρασα ε, του συνεδρίου μας. Θα ήθελα και πάλι να επαναλάβω ότι ήταν η πρώτη φορά που φορείς ε, από ολόκληρο τον κόσμο της Διερμηνίας ε, βρίσκονται στην ίδια αίθουσα και μάλιστα έχουμε εκπροσώπους οργανισμών και πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψηφίων για ένταξη χωρών, εκπροσώπους άλλων μεγάλων γνώσεων του κόσμου ε, και με επικεφαλής των τμήματων διερμηνίας ε, επίσης. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη συνεργασίας και αλληλεπίδρασης όλων αυτών των ανθρώπων και των φορέων. Έχουμε κορυφαίους εμπειρογνώμονες. Είχαμε τη χαρά να ακούσουμε τις συναρπαστικές τους παρουσιάσεις ε, από εμπειρογνώμονες που δεν ήταν κατά ανάγκη και νομίζω ότι μας βοήθησε πολύ η παρουσίαση ε, της προσέγγισης και του πρίσματος ανθρώπων που δεν ε, απολαμβάνουν την δική μας ευτυχία της παραμονής στο ενιδρίο, αλλά για τους οποίους αποτελούμε ερευνητικό θέμα. Πολύ μας ικανοποίησε λοιπόν αυτή η ευκαιρία που είχαμε και ευχαριστώ και την ΑΕΚ που συμμετείχε στην πολύ σημαντική αυτή διά, διάσκεψη και ευχαριστώ θερμά όλους που έκαναν μακρινά ταξίδια γιατί αντιλήφθηκαν τη σημασία που έχει αυτή η πρώτη τέτοιου είδους διάσκεψη Ελπίζω ο κύκλος αυτός να διευρυνθεί, να συνεχιστεί η συνεργασία και η αλληλεπίδρασή μα, γιατί σε ένα παγκοσμιωμένο κόσμο οι ερευνητέ δεν μπορούν να μένουν στη γωνίτσα τους, ούτε τα πανεπιστήμια να μένουν στο δικό τους κόσμο. Αλλά και οι διερμηνείς και οι διεθνεί οργανισμοί επίσης δεν μπορούν να είναι απομονωμένοι. Αναγνωρίζοντας λοιπόν αυτή την αλήθεια, προτείναμε για το συνέδριό μας και μια μεγάλη καινοτομία. Προτείναμε δηλαδή να διευρύνουμε την εικονική εκμάθηση όχι μόνο στα πανεπιστήμια των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι που γίνεται συνήθως με αρκετή επιτυχία από ό,τι ξέρω, δηλαδή ε, δικαστήριο, κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σκεφτήκαμε να βγούμε από το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τεχνικά αυτή τη συνεργασία και με έναν άλλο διεθνή οργανισμό. Και μάλιστα έχουμε ε, τη δεδηλωμένη βούληση και προθυμία δύο τέτοιων διεθνών οργανισμών. Θα εξετάσουμε βέβαια τις τεχνικές παραμέτρους, πάντως σας ευχαριστώ για την προθυμία. Έχουμε το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και το Συμβούλιο της Ευρώπης ε, εκδήλωσαν ενδιαφέρον για ε, τέτοιου είδους τεχνική συνεργασία εικονικής εκμάθησης. Σας ευχαριστώ θερμά γιατί όλο όσο ε, ανοίγουμε τους ορίζοντές μας και κατανοούμε ένα τα, τα προβλήματα του άλλου, τόσο πιο εύκολα θα βρούμε συνέργειες που θα είναι επωφελείς και ευεργετικές για όλους μας. Πέραν όλων αυτών των φορέων, είχαμε στο συνέδριό μας και εκπροσώπους από τις μόνιμες αντιπροσωπείες, από το διπλωματικό σώμα. Γιατί δεν είναι μόνο οι υποψήφιες χώρες που αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα της διερμηνίας. Και άλλες χώρες την αναγνωρίζουν και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων γι' αυτό. Είχαμε ε, διπλωματικές αποστολές από τη Ρωσία, την Κίνα και άλλες χώρες που έδωσαν το παρόν στην εκδήλωσή μας. Ευελπιστώ ότι φεύγοντας από εδώ μετά από ένα ελαφρύ γεύμα που θα απολαύσουμε εκτός της αιθούσης ε, θα κρατήσετε ε, την εικόνα ενός επαγγέλματος ε, εν εξελίξη, ενός δυναμικού επαγγέλματος που αν δεν έχει καταφέρει να, ακόμη να αποκτήσει ένα καθεστώς και μία αναγνώριση α, ποιο, ποιος μπορεί κανείς να ονομάζεται ε, διερμηνέα συνεδριάσεων, συνεδρίων. Νομίζω ότι τουλάχιστον έχει την αναγνώριση όλων όσων χρησιμοποιούν το έργο του διερμηνέα και καταλαβαίνουν ότι αυτό το έργο είναι ένα έργο συνεργασίας, μεταβίβασης μηνυμάτων και διπλωματικής ικανότητας όπως συνέβαινε με τους δραγουμάνους, τους διερμηνείς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και νομίζω ότι οι πρίτενες από τα πανεπιστήμια που ήρθαν στην ε, στο συνέδριο λέγοντας τι θα κάνουμε εμείς σε μια τόσο τεχνική συνεδρίαση, έχουν πια κατανοήσει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, τους προσκάλεσε για την πολύ καλή τους ιατρική σχολή, δεν προσκάλεσε τους Πριτάνης για την πολύ καλή τους νομική σχολή, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τα πανεπιστήμια αυτά γιατί έχουν πολύ καλές σχολές διερμηνίας και πραγματικά είναι της αξίας ε, αυτές οι σχολές και για τα πανεπιστήμια αλλά και για όλους μας. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα θα πρέπει να το διαβιβάσετε και στους ε, αρμοδίους, στις αρμόδιες αρχές. Και ελπίζω ότι στην επόμενη μας ε, διάσκεψη θα έχουμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες επαφής. Πριν περάσουμε λοιπόν στο ελαφρύ γεύμα που σας υποσχέθηκα, θα ήθελα να πω με την αδειά σας ότι αν θα μπορούσα να πω ότι είμαι η μητέρα της ιδέας ε, ε, αυτής της διοργάνωσης, μπορεί εγώ να την εμπνεύστηκα, αλλά η διοργάνωση αυτή θα ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί χωρίς συνεργασία των δύο κυριών που κάθονται δίπλα μου και που πραγματικά αξίζουν το θερμό σας χειροκρότημα. Γιατί οι δύο αυτές κυρίες και οι συνεργάτες τους ε, επεξεργάστηκαν και το περιεχόμενο του προγράμματος, ε, τις προσκλήσεις ε, των ε, ομιλητών, των καλεσμένων, τα ξενοδοχεία, την, τα κοκτέιλ, την, τα γεύματα, το τεχνικό σκέλος. Όλα πέρασαν από τα δικά τους χέρια και δεν ήταν καθόλου εύκολο, σας διαβεβαιώ. Και παρόλο που δεν είναι παρόντες, θα ήθελα να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τον Αντιπρόεδρο, την Επίτροπο και τον Γενικό μας Γραμματέα που μου έδωσαν λευκό επιταγή να διοργανώσω αυτό το συνέδριο. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς μας. Όσοι είχαν την ευκαιρία να μου μιλήσουν, να μου εξέφρασαν τη χαρά τους ε, που συμμετείχαν ε, και έκαναν τη διερμηνία σε μια συνεδρίαση που είχε σαν αντικείμενο το δικό τους έργο. Και πολύ συχνά σε συνεδριάσεις που δεν έχουν εκ των προτέρων τους λόγους, που μερικές φορές δερμηνεύουν σε ακραίες ε, καταστάσεις ε, και υφίστηται ένα κακομεταχείριση, τουλάχιστον το Κοινοβούλιο να γνώρισε το έργο τους. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ τον προγραμματισμό για την επιλογή αυτή τη πολύ καλή ομάδα. Να ευχαριστήσω τον κύριο Λόρι Σουλάγκο και τον τιματάρχη Φίλιπ Τουλκέτα, τους τεχνικούς τη συνεδρίασης. Επίσης τα LSU, τον Φίλιπ Δερίδε και τον Βερνάρ Γκεβάρτ, τη Γενική Διεύθυνση ITEC που μας συνδράμει στα προγράμματά μας ε, τεχνολογικής επέκτασης και διεύρυνσης. Επίσης να ευχαριστήσω τους συνεργάτες όλων των Γενικών Διευθύνσεων που κινητοποιήθηκαν για να γίνει πραγματικότητα αυτό το συνέδριο και η συμμετοχή τους ήταν υποδειγματική και να ευχαριστήσω ιδιαίτερος ολόκληρη την ομάδα της, του τμήματος στήριξης της και όσοι συνεργάζονται με την Ισαβέλα Πατλώτη και το τμήμα επικοινωνίας. Νομίζω ότι είχαμε ένα λαμπρό παράδειγμα τι μπορεί να κάνει η συνεργασία και η συνέργεια και νομίζω ότι είναι πηγή έμπνευση για όλους μας. Πού μπορούμε να φτάσουμε με τέτοια συνεργασία και νομίζω ότι όλοι αξίζουμε ένα θερμό χειροκρότημα. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στο ελαφριό γεύμα και σας εύχομαι όλους καλή επάνωδο. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και ευτυχής που είχα την ευκαιρία να σας δω όλους εδώ. Ευχαριστώ.